Πρόεδρος, να καθίσετε και να ξεκινήσουμε. Κυρία Λίνα, διαδικαστικό. Να πω ότι ε, το ψήφισμα ε, υπό το 54 έχει ικανοποιητικό αριθμό ε, υπογραφών και επομένως μπορεί